Deutsch haben wir Einen schönen guten Morgen. Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που έχετε έρθει όλοι νωρίς νωρίς. Έχουμε ως θέμα της συνεδρίασής μας τη σύσταση σε σώμα της Επιτροπής τη ειδική Επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές ρυθμίσεις τάξε. Φαντάζομαι ότι είσαστε όλοι όσοι έχετε δικαίωμα ψήφου εδώ. Η κυρία Άννα Γκόμες αντικαθιστά την κυρία Ελίζα Φερέρα. Στο ECR ο Άσλι Φόξ αντικαθιστά την ε, κυρία Σουίνμπερν και ο κύριος Μαριά, τον κύριο Δραστροδεύσκη. Στους πράσιρους αντικαθίσταται η κυρία Ζουλή ε, στο EFDD ο κύριος Βάλλη, τον κύριο Πάξας. Το σημειώνω όλο αυτό διότι δεν έρχονται ως αναπληρωματικοί αλλά συμμετέχουν στη συνεδρίαση δυνάμει του καταστατικού. Σήμερα λοιπόν έχουμε μόνο τη σύσταση σε σώμα της Επιτροπής και αφού συσταθεί θα συνεχιστούν οι υπόλοιπε συνεδριάσεις θα καλύψουν τα άλλα θέματα. Προεδρείο μόνο. Λοιπόν, παρακαλώ να έχετε τις κάρτες σας έτοιμες, αν χρειαστούν. Βλέπω, διαπιστώνω ότι έχουμε την απαρτία. όπως προβλέπετε από τον κανονισμό. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Παρακαλώ, πρόκειται για πράξη σύστασης επιτροπής και οφείλουμε να της δώσουμε τη μέγιστη προσοχή μας. Όλοι. Γι' αυτό θα ήθελα λίγο ησυχία. Παρακαλώ λοιπόν τώρα να κάνουμε την επιλογή. Μα αφήστε να τελειώσω την πρότασή μου. Λοιπόν, παρακαλώ να δούμε προτάσεις για τη θέση του Προέδρου. Ο κύριος Μπάλτς έτοιμος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο θα ήθελα να προτείνω τον Αλέλα Μασούρ ω πρόεδρο. Καλώ. Ερωτώ του συναδέλφου αν υπάρχουν άλλε προτάσεις. Όχι. Συμφωνείτε, διαβοή. Τότε λοιπόν ε, διαπιστώνουμε την εκλογή του Αλέλα Μασούρ ομόφωνα στη θέση του Πρόεδρου και του παραδίδουμε την καθοδήγηση της συνεδρίασης. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον Μάρκους Φέρμπερ, αλλά θα ήθελα και να τον μεμφθώ λίγο, γιατί θα έπρεπε δυνάμει της διαδικασίας να εξασφαλίσει και την ε, συνένεση του υποψηφίου προτινομένου. Αλλά, εν πάση φαντάζομαι ότι μέσα στο γενικό ενθουσιασμό και τη χαρά το θεώρησε δεδομένο. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την τιμή που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Προσδιορισμός των λοιπόν μελών του Προεδρείου. Η διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει ότι πρέπει να υπάρχουν τρεις αντιπρόεδροι και έτσι σας καλώ να ε, ψηφίσουμε έναν πρώτο αντιπρόεδρο καταρχάς. Υπάρχει υποψήφιος ή πρόταση. Ο κύριο Μέσσερ Σμιτ. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρου τη Ομάδα Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Μπέρντ Λούκε ω υποψήφιο. Ε, ε, Κύριε Μπέρντ Λούκε, έχετε νομίζω ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το από τις διατάξεις περί οικονομικών συμφερόντων, δέχεστε την υποψηφιότητα. Πολύ καλά. Λοιπόν, θα πρότεινα διαβοής να εκλέξουμε τον κύριο Λούκη. Κυρία Γκουλάχ, πρόεδρε εκ μέρους της Άλντε, εγώ θέλω ψηφοφορία, πρόεδρε. Καλώς. Τότε διανατάσσεως της χειρός, παρακαλώ, υπέρ της ψηφοφορίας του κυρίου Λούκε. Tous sur les nominations Μπορεί να είναι μυστικές οι ψηφοφορίες, Πρόεδρε, και θα ήθελα να είναι μυστική. Μπορεί να είναι μυστική η ψηφοφορία αν το ζητήσουν 8 βουλευτές. σαν Δεν το ζητούν 8 βουλευτές και έτσι διανατάσσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Έξι και σας ευχαριστώ. Άρα ο κύριος Λούκε εκλέγεται πρώτος αντιπρόεδρος και τον καλό να αναλάβει τα καθήκοντά του. Θέση δεύτερο αντιπρόεδρο. Υπάρχει πρόταση για υποψηφιότητα. Παρακαλώ. Κύριε Ντιμάζιο. η Γκουέντζιελ ήθελε να προτείνει τη Μάρισα Ματίας. Σας ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν. Όχι. Κυρία Ματέας έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Δέχεστε την υποψηφιότητα, κυρία Ματέας. Μάλιστα. Τότε λοιπόν προτείνω ανατάσσω στις κυρώσεις, αν συμφωνώ όλοι επί της αρχής, να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Αντιρρήσεις δεν βλέπω. Αποχές δεν βλέπω. Συγχαρητήρια, κυρία Ματίας. Madame, prenez votre Παρακαλώ, περάστε στο Προεδρείο. Και τέλει, για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Κύριε Γκίγκολτ. Εξ ονόματος ε, των Πρασίνων θα ήθελα να προτείνω την κυρία Εύα Ζολή για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ζολή δεν παρίσταται. Βρίσκεται σε αποστολή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αλοδαπή. Έχει κάνει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και επίσης μας έχει ενημερώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στην υποψηφιότητα. Μπορούμε λοιπόν και τη δική της υποψηφιότητα να την πραγματοποιήσουμε διανατάσεως ή διαβοής, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Καλώς. Υπέρ παρακαλώ. Κάτα. Εποχές. Εκλέγεται λοιπόν και η κυρία Ζολή και τη συγχαίρουμε θα, την, θα τις φτάσουν μέχρι το Αφγανιστάν τα χειροκροτήματά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Δεν θα σας κρατήσω παραπάνω. Μόνο δύο σημεία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχουμε μια αποστολή πολύ σημαντική. Θα είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι στην εξέταση των μέσων μαζικής ενημερώσεις και της κοινή γνώμης. Έχουμε υποχρέωση αποτελέσματος λοιπόν και δι αποτελέσματος ταχύτατο. Η διάσκεψη των Προέδρων θέσπισε με εντολή εξάμηνη την εντολή μας, την Επιτροπή μας. Ε, πρέπει και εμείς να αξιοποιήσουμε αυτή την ορμή που μας δίνει η συγκυρία. Λόγω των αποκαλύψεων που εμφανίστηκαν στον τύπο. Και έτσι να θέσουμε τέρμα σε μία σειρά πρακτικών οι οποίες είναι σαφώς αμφισβητήσιμες. Είναι ένα θέμα λοιπόν αυτό για το οποίο και δεν είναι συνηθισμένο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ευρύτατη συνένεση, ανεξαρτήτως πολιτικής οικογένειας, ε, χώρας προελεύσεως ή και θέσεως απέναντι στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, συμμεριζόμαστε τη βούληση να εξασφαλίσουμε πολιτική δικαιοσύνη, διαφάνεια, δικαιοσύνη και να θέσουμε τέρμα σε καταχρηστικές πρακτικές. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τις βέλτιστες συνθήκες και τη βέλτιστη διάθεση. Διαπιστώνω ότι η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Τάξε είναι ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Μέλος της, ε, μέλος της Επιτροπής μας άλλωστε είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα μεριμνήσουμε λοιπόν με τον συνάδελφο αλλά και με όλους τους άλλους βουλευτές σε κάθε δραστηριότητά μας, να μην μπαίνει σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής των Οικονομικών η Επιτροπή Τάξε και τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν να τα εξετάζουμε με πνεύμα επικοδομητικό, χωρίς επικάλυψη και σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας. Κοιτάξτε, η πρόθεσή μου δεν ήταν να αρχίσω συζήτηση, αλλά βλέπω ότι ο κύριος Λάμπερτς μου ζητάει διαδικαστικό. Ε, Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι διαδικαστικό. Μια και είχα την πρωτοβουλία που οδήγησε, αν θέλετε, στη σύσταση αυτής της Επιτροπής, θα ήθελα να κάνω μία δήλωση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω το γεγονός ότι στο μυαλό μας πάντα ήταν σαφές ότι ο στόχος των εργασιών που θα ξεκινήσουμε είναι ένας στόχος που επιδιώκει να αλλάξει τις πρακτικές. Κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να λιντσάρουμε δημόσια είτε χώρες είτε επιχειρήσεις ή άτομα. Θέλουμε να αμφισβητήσουμε πολλές πρακτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός και αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία για τη σύσταση αυτής της ειδικής επιτροπής είναι ακριβώς να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη δικαιοσύνη. Αυτό είναι η λέξη, η έννοια κλειδί. Θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσουμε γρήγορα, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορμή που έχει δημιουργηθεί και αν αποδειχθεί ότι δεν μπορούμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να προτείνουμε στην διάσκεψη των Προέδρων μία παράταση πρέπει να καταβάλουμε τις βέλτιστες προσπάθειες για να καταλήξουμε το ταχύτερο. Πρόκειται για ένα ευρύ θέμα, η εντολή που μας δόθηκε είναι και αυτή ευρεία, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε βάθος και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους όσων είχαν την πρωτοβουλία, δεν είναι θέμα να αντιπαρατεθούμε μεταξύ μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά αυτής της Επιτροπής έχει λήξει σαν θέμα συζήτησης. Τώρα θέλουμε να εξελίξουμε τις πρακτικές σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη δήλωση, λέει ο Πρόεδρος. Όσον αφορά την επιθυμητή διάρκεια των εργασιών μας, η, η εμπειρία μου δείχνει ότι Όσον αφορά την πολιτική εργασία, ο φυσικός νόμος του Απογκαντρό Λεπέρ έχει εφαρμογή. Δηλαδή η εργασία καταλαμβάνει όλο τον χρόνο που έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε. Αν αποφασίσουμε λοιπόν να ε, ε, εξετάσουμε ένα θέμα για δύο χρόνια, θα το χρειαστούμε δύο χρόνια. Αν αποφασίσουμε να το ε, αντιμετωπίσουμε μέσα σε δύο ώρε. θα το ε, οριστικοποιήσουμε σε δύο ώρε. Έξι μήνε, έξι μήνε. Λοιπόν, ε, συμμερίζομαι την άποψή σα. Ο κύριο Τόιρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια καταρχά για την εκλογή σα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η προστασία του, των πνευματικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να επισημάνω ότι εγώ ήμουν εκείνο ο οποίο το Σεπτέμβριο σε μια συνεδρία τη Επιτροπή των Οικονομικών και Νομισματικών ε, Θεμάτων εκ μέρου τη ομάδα Άλντε είχα ζητήσει να υπάρξει μια <clears throat> επιτροπή για τη διερεύνηση των θεμάτων, μια ειδική επιτροπή ε, για τι φορολογικέ ρυθμίσει τύπου tax rulings. Χαίρομαι λοιπόν που συνίσταται αυτή η επιτροπή και χαίρομαι που μπορέσαμε να συμβάλλουμε στο να μπει στο θεματολόγιο, στη δουλειά του Κοινοβουλίου η εξέταση των θεμάτων αυτών. Θέλουμε, πιστεύω, να πούμε ότι, ήταν πολύ, ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε προχωρήσει ταχύτατα στην θέσπιση αυτής της ειδική Επιτροπής, γιατί απεδείχθη ότι δεν χρειάζεται να χάσουμε τόσο χρόνο. Είναι ο καταλληλότερος τρόπος να διερευνηθούν τα ζητήματα της, ε, φορολογικής, της επιθετικής φορολογικής ε, πολιτικής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των προκατακτικών ρυθμίσεων. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, να μην χάσουμε την ορμή που μας δίνει αυτή η συγκυρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προχωρήσει και να πάρει την πρωτοκαθεδρία στην εξέταση, στην διερεύνηση καλύτερα των θεμάτων αυτών. Θέλουμε να δουλεύουμε σωστά για τα θέματα αυτά και το μόνο που έχω να πω είναι ότι καλό γιατί η διάσκεψη των Προέδρων μίλησε για μια ειδική επιτροπή, επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές ε, ρυθμίσεις κτλ. Θέλω λοιπόν να πω, μια και ο κύριος Μέθερ Σμιτ και ο υποφαινόμενος ως ε, συνεισηγητές ε, στις προτάσεις που έχουμε αναλάβει να διατυπώσουμε, έχουμε την εντολή αυτή, ε, θα πρέπει να επισκεφθούμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και άλλες ε, χώρε. Έχουμε μια ειδική λοιπόν επιτροπή τώρα, με την οποία δεν θα μπορέσουμε εμείς να αναλάβουμε τις ε, εκθέσεις, τις εισηγήσεις και άρα θα ήθελα στηριζόμενοι στις εισηγήσεις που έχουμε συντάξει με τον κύριο Μέσσαρσμιτ μαζί να προχωρήσουμε και να αναπτύξουμε το έργο. κύριος Λόγος. Σημειώνω λοιπόν ότι είστε πανέτοιμος να εργαστείτε και ότι έχετε ήδη πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για να επιταχύνετε τα αποτελέσματα. Ο κύριος Τιέρη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Η Σωσιαστική ομάδα χαίρεται για τη συγκρότηση αυτής της επιτροφής. Χαιρόμαστε που πολλοί θεωρούνται πρωτεργάτες της Επιτροπής αυτής. Θετικό αυτό, επειδή δείχνει ότι την... έτσι στερνίζονται όλοι αυτή την Επιτροπή, όλες οι πολιτικές ομάδες. Ελπίζουμε λοιπόν να βοηθήσουμε στις εργασίες μας και χαιρόμαστε που συμβάλαμε και εμείς στην ε, ανέβρεση λύσης σχετικά με τη συγκρότηση αυτής της ομάδας ως πρόταση στην διάσκεψη των Προέδρων. Να σας πω ότι εκτίμησα πολύ την εισαγωγική σας ομιλία και την βούληση για στενή συνεργασία και την ε, νομοθετική πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει η Επιτροπή μας σε λίγο. Έχουμε εδώ την συγγήτρια δίπλα μου και νομίζω ότι η διάκριση των ρόλων και η συνεργασία μπορούν να αποβούν πολύ επωφελείς στα πλαίσια της θητείας αυτής της Επιτροπής μας στην εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων βεβαίω που αφορούν τις φορολογικέ ρυθμίσει. Λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω και τι υποχρεώσει που θέτουν οι συνθήκε, με τι οποίε όμω δεν υπάρχει άμεση σύνδεση των φορολογικών ρυθμίσεων. Με χαρά λοιπόν θα βοηθήσουμε στην δεξαγωγή των εργασιών και χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να υποβάλει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου, όχι μόνο για να κάνουμε μια διάγνωση των δεινών που μαστίζουν την Ευρώπη, αλλά για να βρεθεί και η σωστή θεραπεία. Καλή δουλειά σε όλους μας. Ε, Ευχαριστώ, Ρομπέρτο Μπούρκο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχάς, από πλευράς μου, αλλά και ολόκληρου του ΕΛΚ, ασφαλώς ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την ανάληψη τη θέση του Προέδρου της νέας αυτής ειδικής επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρο, όπως τονίσατε και εσείς, στους επόμενους μήνες όλοι και ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας να φροντίσουμε να συνεργαστούμε καλά. Θέλουμε κι εμείς στους επόμενους μήνες να προκύψουν καλά αποτελέσματα. Ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη άλλωστε μίλησε για τη στενή συνεργασία με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό πιστεύω κι εγώ. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα αντίστοιχα με αυτά ε, με, την με το νομοθετικό ψήφισμα και ως εκ τούτου νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συνεργαστούν στενά οι δύο επιτροπές, η Ειδική Επιτροπή μας και η Οικονομική και Νομισματική. Έξι μήνες καλή συνεργασία πιστεύω ότι μας περιμένουν. Περιμένω με αδμονία να δω πώς θα προχωρήσει η δουλειά αυτή. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα και νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να πω πια από πλευράς μας είναι ότι μπορεί να ξεκινήσει η δουλειά. Ευχαριστώ αγαπητέ Μπορουκάρτ. Φάβιο Πρόεδρε, για άλλη μια φορά και εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή σας και την εκλογή των αντιπροέδρων. Πρέπει να πω ότι με ξαφνιάζει αυτός ο ε, νεόκοπος ενθουσιασμός του Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση των ε, καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών. Πάντως το χαίρομαι και καλό θα είναι να υπενθυμίσουμε ανεξαρτήτως του ποιος διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα, ότι η ομάδα της Γκουέ ήταν εκείνη η οποία ή μη τι άλλο ε, ε, υποδάβλησε αυτόν τον ενθουσιασμό για την καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών. Και θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερος ότι καθήκον μας είναι μαζί, να, να ακολουθήσουμε βεβαίως το ευρωπαϊκό δίκαιο, με βάση αυτό να κρίνουμε, αυτό θα πράξουμε άλλωστε, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση και διαφάνεια όσον αφορά τα έγγραφα. Αυτό ισχύει και ε, με την επισήμανση ότι ένα από τα προβλήματα που είχαμε και εμείς αλλά και η ομάδα των Πρασίνων και άλλοι που μας υποστήριξαν ήταν όταν ζητούσαμε να έχουμε τα σχετικά έγγραφα ε, πέφταμε πάνω σε κλειστές θύρες σε σχέση με, τα, με τις αποφάσεις και τα έγγραφα που αφορούν τη φορολογική πολιτική των κρατών. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε μέγιστη διαφάνεια ως προς την διάθεση των εγγράφων Χαίρομαι που ο Πρόεδρος ε, μίλησε για την ορμή που μας δίνει η τωρινή συγκυρία, η στιγμή, η ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Βλέπω ότι όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό ξεκινούν. Ελπίζω ο ενθουσιασμός να κρατήσει και κατά το πέρας του εξαμήνου να είναι ακόμη ορατός. Εάν χρειαστεί όμως θα πρέπει να ζητήσουμε την παράταση της εντολής μας εφόσον δεν έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας μέχρι τότε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφο, ο κύριο Φόξ είναι ο τελευταίος ομιλητή. Καλημέρα κύριε Λαμασούρ, συγχαρητήρια για την εκλογή σα. Η ομάδα μας προσλέπει σε συνεργασία με την Επιτροπή αυτή και αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, διακόπτει ο μιλητής γιατί κάποιοι δίπλα μιλάνε, περιμένω ο συνάδελφο να τελειώσει εδώ με το τηλεφώνημα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι στη δουλειά μα, τότε να θυμόμαστε εμεί τα μέλη ότι η φορολογική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών μελών. Πολλοί από εμά εδώ θεωρούν ότι ο ανταγωνισμός ο φορολογικό μεταξύ χωρών μελών είναι κάτι καλό και κάνει το κράτος έντιμο, ειλικρινές, ώστε να μην παίρνει μεγάλο κομμάτι των εισοδημάτων των πολιτών. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξουμε το βαθμό με τον οποίο οι χωρισμένοι χρησιμοποιούν τις φορολογικές πολιτικές για παράνομες κρατικές επιδοτήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε πώς οι χώρες έχουν χρησιμοποιήσει αυτές τις φορολογικές πολιτικές για αυτούς τους σκοπούς. Αν θέλετε να έχουμε περισσότερη λοιπόν Ευρώπη, Ευρώπη που θα πρέπει να καθορίζει την φορολογική πολιτική των μελών, τότε θα αγνοηθούμε από το Συμβούλιο. Θα προτείνω λοιπόν στα μέλη να κάνουμε κάτι επικοδομητικό και να επικεντρωθούμε στενά σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποδεχτεί χρήσιμο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε από αυτού. Αγαπητέ συνάδελφοι, σα ευχαριστώ. Τελευταίο σχόλιο από τον πρόεδρο Βολφ Κερή. Παρακαλώ μην πάρετε πολύ χρόνο, διότι σε δύο λεπτά θα έχετε να προεδρεύσετε στη διπλανή αίθουσα. Ναι, θα δώσουμε ένα αντίγραφο στον συνάδελφο Φόξ των ευρωπαϊκών συνθήκων που αναφέρονται όλε οι διατάξει τη Ένωση σε σχέση με τα φορολογικά θέματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα διανύμουμε επίση όλα τα μέλη την εντολή που μας έδωσε η διάσκεψη των Προέδρων που αναφέρεται στην πολιτική ανταγωνισμού πράγματι. Πριν φύγετε αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ε, που ο κύριος Δαμασί ε, αναφέρεται στον συλλογικό ενθουσιασμό που δεν με εντυπωσιάζει. Η πατρότητα αυτής της πρωτοβουλίας ανήκει σε πολλούς, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους. Αλλά η νίκη πάντα έχει πολλούς πατέρες, η ήττα είναι ορφανό. Έχουμε λοιπόν 45 πατέρες για τη νίκη μας, ελπίζω, σε 6 μήνες ή λίγο παραπάνω η επόμενη μας συνεδρίαση όπου θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε προσδιορίζοντας τον εισηγητή κτλ. θα γίνει στις 9 Μαρτίου στο Στρασβούργο αμέσως μετά τη συνεδρίαση ΕΚΟΝ σε 9 το βράδυ. Είναι λίγο αργά αλλά θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Λύε τη συνεδρίαση.